Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Κυρίσω την έναρξη των εργασιών μας. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ε, ιού του AIDS από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι μετά από τη δήλωση της Επιτροπής θα ακολουθήσει ένας γύρος ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και ότι δεν θα διεξαχθεί διαδικασία Catch the Eye. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ντάλι εξ ονόματος της Επιτροπής να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι σήμερα. Sorry. Σήμερα το βράδυ υπομιλητής ε, πρόκειται για λαθάκι. Στην Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για το ψήφισμα σχετικά με την ανταπόκριση ε, για την καταπολέμηση του AIDS που θα εγκριθεί σήμερα. Σημεριζόμαστε την ανησυχία και τη δέσμευση που έχετε αναλάβει για να βελτιώσετε τη ζωή όλων των οροθετικών και όσων πάσχουν από AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψήφισμα είναι ένα ηχηρό και επίκαιρο μήνυμα που τονίζει ότι εδώ και 30 χρόνια καταπολεμούμε την νόσο και παρόλα αυτά είναι πήγον το θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. 25.000 άνθρωποι μολύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φέτο και πάνω από 100.000 νέα κρούσματα αναφέρθηκαν στι ε, στις ανατολικές γειτονικές χώρες. Έχουμε αναλάβει δέσμευση για καθολική πρόσβαση στην πρόληψη, στην περίθαλψη ούτω ώστε ε, να επιτύχουμε μέχρι το 2015 τους στόχου της χιλιετίας. Θα ήθελα να σα καθησυχάσω λέγοντα ε, ότι συνιστά ακόμη προτεραιότητα, υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταπολέμηση του AIDS. Πριν από δύο χρόνια είχαμε υιοθετήσει ένα σχέδιο δράση για την καταπολέμηση τη νόσου εντό τη Ένωση και στι γειτονικέ χώρε έκτοτε. Η Επιτροπή υποστήριξε διάφορε πρωτοβουλίε σε αυτό το τομέα. Τα κράτη-μέλη και οι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετείχαν στα ανεπτυξιακά προγράμματα και στις διμερείς συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Ε, όντως ε, υπάρχουν ε, τεκμήριο ότι με γενικευμένη πρόσβαση στην πρόληψη και στην περίθαλψη και καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης βρίσκονται στον πυρήνα της εκστρατείας καταπολέμησης της νόσου. Επίσης, έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ώστε να συντονίσουμε τις διάφορες επιμέρους πολιτικές, όπως παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, είναι την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Καταπολέμηση του ΟΗΤΣ. Πριν από δύο χρόνια το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψηφίστηκε, αλλά παραμένει ενισχύ και θα καταθέσουμε αναφορέ στι αρχέ του 2012 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματο. Ε, Κυρίω ε, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που ζούμε, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη σημασία της καταπολέμησης της νόσου. Θα συνεχίσουμε να διαδραματίσουμε, να διαδραματίσουμε ενεργό και δραστήριο ρόλο σε αυτό το τομέα και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να τονίσω ότι βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας ε, ω προ τη νέα πολιτική υγείας που σύντομα θα σχολιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε Ντάλη. Θα περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Φρανσουάζ Γκροστέτ εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης ε, του AIDS. Πολύ σημαντικό θέμα για το Κοινοβούλιο μας και πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο μας να εκπονήσει το ψήφισμα αυτό, το οποίο θα πρέπει να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα, γιατί ναι, μεν υποχωρεί κάπως ε, η ασθένεια, ε, μειώνεται όμως και η προβολή της και δεν πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειες. Εξακολουθεί να αποτελεί μάστιγα. Πάνω από 12 εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 25 ετών, 500.000 στην Ευρώπη πλήττονται από τον ιό αυτό. Γι' αυτό πρέπει να ενώσουμε τις πολιτικές μας δυνάμεις. Η Επιτροπή, το είπε και ο Επίτροπος Νταλή, υιοθέτησε ένα πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση του ιού για την περίοδο 2009-2013. Είναι πολύ σημαντικό τώρα που είμαστε στα μέσα του δρόμου να μπορέσουμε να κάνουμε μια εκτίμηση της κατάστασης και να δούμε τι πετύχαμε. Ποια είναι η διάγνωση. Κάθε χρόνο πάνω από 50.000 νέες περιπτώσεις οροθετικών διαπιστώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γείτονε χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 30% οι οροθετικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν ότι είναι μολυσμένοι από τον ιό και σε άλλες χώρες φτάνει το 70%. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τους πολιτικούς ηθήνοντες όπως είμαστε εμείς. Οι μισοί από τους οροθετικούς εξακολουθούν να λαμβάνουν θεραπεία πολύ αργά και φτάνουν σε στάδια μόλυνσης πολύ προχωρημένα πριν καν να διαγνωστεί η περίπτωσή τους. Επιπλέον, πρόσφατα αποδείχτηκε ότι ένας οροθετικός ο οποίος παίρνει αντιρετροϊκά φάρμακα πριν ε, ε, αρχίσει να επιδεινώνεται η υγεία του μπορεί να μειώσει κατά 96% τις πιθανότητες να μολύνει του συντρόφου του. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει τις προσπάθειές της, ώστε να αποδώσουν οι επενδύσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, να φροντίσουμε για την ενημέρωση, να φροντίσουμε για τον έλεγχο, να φροντίσουμε αδιάκοπα ε, να συνεχίσουν να λειτουργούν τα δίκτυα εκείνα τα οποία βοηθούν την καταπολέμηση της μάστιγας αυτής. Και επίσης να ενημερώσουμε και να διαδώσουμε τις καλές πρακτικές. Για παράδειγμα, να γίνονται πολύ εύκολα ε, τα τεστ η αιματολογική έλεγχη στους πολίτες. Αν είναι κάτι συνηθισμένο και διαδεδομένο στις κοινωνίες μας, θα είναι πιο εύκολο καθένας από εμά να πηγαίνει να ελέγχεται και να γνωρίζει κατά πόσο έχει μολυνθεί ή όχι. Να λοιπόν τι δουλειά πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην σταματήσουμε τις προσπάθειες, αλλά να τις συνεχίσουμε για να καταφέρουμε να αντιπολιμήσουμε τον ιό του AIDS. Ευχαριστώ την κυρία Γκροστέτ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Τσάιλντερς εν ονόματι των σοσιαλιστών για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, ε, ε, το AIDS ορτάζει τα 30 χρόνια από τον εντοπισμό της πρώτης, ε, του πρώτου περιστατικού και είναι η ευκαιρία να θυμηθούμε αυτούς οι οποίοι πέθαναν και ε, να θυμηθούμε το σημαντικό αυτό ιό και γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συμβάλλει ή στην καταπολέμηση του ιού στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις γειτονικές χώρες διότι διαπιστώνουμε ότι 30% των ατόμων που ε, ε, είναι φορείς του ιού δεν το γνωρίζουν και γι' αυτό ε, πρέπει κανείς να ενημερώσει τους νέους, τους φυλακισμένους, τους εργαζόμενους στον τομέα του σεξ διότι έχουμε επενδύσει Πόρου ε, πόρους για ε, το, την ομάδα υψηλού κινδύνου σε κλινικές, ε, σε ναρκωμανείς και πολλές δοκιμές έχουν γίνει σε κλινικά εργαστήρια και αποτελούν μέρος του προγράμματος αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές νέες διαγνώσεις και πρέπει η κοινωνία να συμβάλλει εις ε, την διάγνωση και τον εντονισμό, να εντείνουμε την προσπάθεια και ιδίως να στηρίξουμε μία προσέγγιση που να βασίζεται στην κοινωνία για να αποφευθεί το στίγμα και η διάγρυση. Οι ασθενείς από AIDS πρέπει να ε, την χάνουν ίσης μεταχείρισης και ε, η μελέτη του ΟΗΕ το 2010 διεπίστωσε ότι υπάρχει πολύ ανητική στάση έναντι αυτών των ασθενών οι οποίοι έχαναν τη δουλειά τους, αποκλείονταν από τις οικογενειακές ε, εργασίες και ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο εχθρός μας είναι ο ιός και όχι οι φορείς. Θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις ε, να αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό στα πλαίσια της αποκατάστασης σεξουαλικής υγείας να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και να ενισχύσουμε τα ε, δικαιώματα των γυναικών. Ε, λυπούμε, ε, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμη αναπτύξει μία στρατηγική και οι περισσότεροι σε επίπεδο εθνικό και διεθνές πρέπει να συμβάλλουν και ιδίω ο συνάδελφος Μάικελ Κάσου που έχει εργαστεί τόσο σκληρά επί αυτού του θέματος για τόσο χρόνο. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Παρβάνομα, εξ ονόματος της ομάδας των Φιλελευθέρων, για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Thank you, Madam President. Mr. Commissioner, dear colleagues. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Τόσα χρόνια μετά τους αγώνες καταπολέμησης του AIDS στις χώρες μας αλλά και στις γείτονες χώρες, Πρέπει να ομολογήσουμε ότι είμαστε μακριά από το στόχο που είχαμε βάλει να έχουμε μηδέν μολύνσεις από το AIDS. Άρα χρειάζεται να επιτεθεί επιπλέον πρόοδος όταν μιλάμε για την πρόληψη, για την έγκαιρη διάγνωση, για τη σωστή θεραπεία. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ξεχνιέται μερικές φορές ε, η ασθένεια στα μυαλά των ε, πολιτικά εθνόντων. Όμως μετά από τόσα χρόνια πρέπει να συνεχίσουμε να υπογραμμίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η ενημέρωση του κόσμου και η ανάγκη πολιτικών που προλαμβάνουν τη μόλυνση από το AIDS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τη δέσμευσή της. Κύριε Επίτροπε, χαιρόμαστε για τη δέσμευση που μας ανέφερε ο Επίτροπος, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τον αγώνα κατά του AIDS. Ελπίζουμε όμως ότι θα ξεκαθαρίσετε στα κράτη-μέλη ότι δεν φτάνει μια στρατηγική στα χαρτιά. Ακόμα και τώρα που είμαστε σε οικονομική κρίση, πρέπει τα αντίστοιχα προγράμματα καταπολέμησης του AIDS να τίθεται σε εφαρμογή. Να δούμε την πραγματικότητα, να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες δεν έχουμε περιθώρια για ταμπού. Είναι πολύ βασικό τα κράτη-μέλη να φροντίσουν όλα τα εθνικά προγράμματα καταπολέμησης του AIDS και όλα τα προγράμματα ενημέρωση ε, ε, σχετικά με το AIDS να τεθούν σε εφαρμογή. Σήμερα θα ψηφίσουμε ένα ψήφισμα το οποίο στηρίζεται από όλε τι πολιτικέ ομάδε στην Επιτροπή περιβάλλοντο. Ναι, υπάρχουν ε, ομάδε πιο ευάλωτε νέοι, ομοφιλόφιλοι, ε, οι χρήστες ε, ναρκωτικών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κατάλληλες στρατηγικές. Οι ομάδες αυτές είναι ευάλωτες και από, άλλες, ε, από άλλα προβλήματα, αποκλεισμός, κοινωνικός αποκλεισμός, από τα οποία επίση αποφέρουν. Δεν πρέπει να αρνιόμαστε την ύπαρξη των ατόμων αυτών ή να αρνιόμαστε να μιλάμε για εκστρατείε κατά των διακρίσεων. Όχι, είναι και αυτά μέρος της καταπολέμησης του AIDS. Ελπίζω ότι όλοι οι βουλευτές εδώ δεν θα δούνε ιδεολογικά το θέμα και θα υποστηρίξουν το ψήφισμα. Είναι μια ευκαιρία να επενθυμίσουμε ότι επιμένουμε στον αγώνα αυτό, ότι είμαστε δεσμευμένοι για την καταπολέμηση του AIDS στην Ευρώπη και την εξαφάνισή του. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροτ Μπέρεντ έχει σηκώσει μπλε κάρτα. Θα ήθελε να κάνει μια παρέμβαση. Δέχεστε την μπλε κάρτα. If you accept Δέχεστε την μπλε κάρτα. Η κυρία Ροτ θέλει να σας θέσει ε, ένα ερώτημα. Κυρία Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Παρβάνοβα το εξή. Συμφωνείτε μαζί μου. Εντάξει, αληθεύει ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια στον προπολογισμό τη Ένωση ε, για να έχουμε προγράμματα επιμόρφωση, ενημέρωση, ε, ε, καταπολέμηση του AIDS. Πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη παραμελούν τα καθήκοντά του σε σχέση με την ασθένεια. Η κυρία Τσάλλας ε, αναφέρθηκε σε αριθμητικά στοιχεία που όλοι γνωρίζουμε ότι αληθεύουν. Μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να μας δείξουν πόσα χρήματα ε, δαπανούν για την εκστρατεία ενημέρωση ε, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για την εκρίζωση του νόσου. Πρέπει να ζητήσουμε ίσω από την επερχόμενη Προεδρία τη Δανική να κάνει κάποια βήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ροτ Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να υλοποιήσουμε την πολιτική. Το σημαντικό είναι να λειτουργεί αποτελεσματικά η πολιτική και εδώ πέρα χρησιμοποιούμε τις ευκαιρίες που έχουμε για την καινοτομία, για τις εταιρικέ σχέσεις. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για την αποτίμηση της κατάστασης σε σχέση με την νόσο. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλά αποτελέσματα, γιατί είναι κέρια σημασία να επικρατεί η διαφάνεια σε σχέση με τι ροέ κονδυλίων που διοχετεύονται για την υλοποίηση κάποιων προτεραιοτήτων και να δούμε αυτά τα κονδύλια, ποια προστιθέμενη αξία έχουν σε σχέση με αυτή τη διαδικασία και την εφαρμογή των πολιτικών. Διότι εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε ανέκαθεν επίγνωση τη πίεση που ασκείται προ όλε τι κατευθύνσει για πράγματα που δεν είναι σημαντικά για την Ευρώπη ούτε για, τις πολι... για τους πολίτες. Ε, για κάποιους από τους λομπίστες ε, είναι σημαντικό βέβαια το θέμα. κάνουμε κάτι που θα είναι υποφελέ για όλους τους πολίτες. Ευχαριστούμε κυρία Παρβάνοβα. Παρακαλέσω την κυρία Γιάννα Κουδάκη εξ των Ευρωπαίων Συντηρητικών να πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα θυμόμαστε με μεγάλη θλίψη τις πολλές αθώες ζωές οι οποίες χάθηκαν μέσω αυτής της τρομερής ασθενείας. Δεν βλέπουμε μείωση στον αριθμό των νέων μολύνσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτό δεν επαρκεί. Είναι μια επιδημία η οποία πλήττει όλα τα κράτη-μέλη και έχουμε ευθύνες έναντι αυτών οι οποίοι ζουν με το, και φέρουν τον ιό. Εξού και σήμερα είναι η μέρα για την αντιμετώπιση του AIDS από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση για την έρευνα για να ευρεθεί ένα εμβόλιο. Γνωρίζουμε μία ασθένεια η οποία δεν γνωρίζει ούτε σύνορα, ούτε ηλικία, ούτε φίλο Αλλά είναι μία ασθένεια την οποία μπορούμε να ελέγξουμε, ιδίω μέσω των εξετάσεων και ελπίζουμε ότι κάποια μέρα θα βρούμε και μία θεραπεία. Μέχρι στιγμής πρέπει να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση, να ενισχύσουμε τις εργασίες μας και ε, να συμμεριζόμαστε τα απορίσματα των ερευνών μας. Γι' αυτό και η πολιτική μου ομάδα ε, παραστέκεται σε όλες τις οικογένειες και όλους που θυμούνται τα άτομα που υπέκυψαν στο AIDS για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών οι οποίοι ζουν με τον ιό και ε, να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε δεσμευμένοι να καταπολεμήσουμε ε, την ασθένεια. Του χάσει εξ της ομάδας των Για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους οι οποίοι συνεισέφεραν στην ε, εκπόνηση του ψηφίσματος αυτού. Έχουμε ένα κοινό στόχο και ο κοινός μας αυτός στόχος είναι να μειωθούν οι περιπτώσεις ε, μόλυνσης από το AIDS στην Ευρώπη. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λάβετε υπόψη σα και τις γείτονες χώρες, τότε έχουμε πάνω από 100.000 νέες περιπτώσεις το χρόνο. Και είναι και μια ασθένεια η οποία θα μπορούσε να αποφευθεί πλήρως. Και ξέρουμε πώς. Ξέρουμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη διάδοση του AIDS. Οι νέες περιπτώσεις μόλυνσης από το AIDS θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν το έχουμε καταφέρει. Στη Νότια Αφρική πρόσφατα είδα ε, μια διαφήμιση στην τηλεόραση. Εκεί ο Νέλσον Μαντέλα έλεγε «Αγαπάμε τα παιδιά μας». Γι' αυτό και θα πρέπει να μιλήσουμε μαζί τους για το σεξ. Θέλω να πω με αυτό ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν πώς διαδίδεται το έτσι, πώς μπορεί να μολυνθούν από τον ιό και πώς μπορούν να το αποφύγουν, όπως επίσης πόσο μεγάλη σημασία έχει η χρήση των προφυλακτικών. Στη χώρα μου, τη Φιλανδία, η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο είναι κάτι που επιτρέπει να συζητιώνται τα θέματα που έχουν να κάνουν με το σεξ και είναι ένας αρκετά αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία απορρέουν από μια συγκεκριμένη σεξουαλική συμπεριφορά. Η ε, διάδοση δηλαδή των σεξουαλικά μεταδεδομένων ασθενειών, AIDS, αλλά και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Η Φροντίδα για την υγεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί συνάδελφοι εδώ αναφέρθηκαν ειδικά στις γυναίκες. Σύμφωνα με τις ε, στατιστικές, το 45% των νέων μολύνσεων αφορά νέες γυναίκες κάτω των 25. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι και θέμα φύλου το AIDS. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο οι γυναίκες είναι ενημερωμένες για την αναγκαιότητα χρήσης προφυλακτικού και αν ε, το ζητούν κάθε φορά. Ξεκάθαρα λοιπόν ε, μπορούμε να πούμε ότι όσοι δεν είναι ενημερωμένοι για το ότι είναι οροθετικοί ε, κινδυνεύουν περισσότερο να κολλήσουν τους συντρόφους τους και να περάσουν επίσης και τον ιό στα ίδια τους τα παιδιά. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι η φροντίδα για τους ασθενείς του AIDS. Πρέπει να αποφύγουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και χρειάζονται στόχοι μετρήσιμοι, παρακαλώ. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία ε, Μαρίζα Ματίας, ε, εξ ονόματος της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Είμαστε εδώ σήμερα όλες ε, και όλοι ενωμένοι γύρω από ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου κάνοντας πολύ σημαντικά αιτήματα για τις παρεμβάσεις στον τομέα της καταπολέμησης του AIDS. Είναι η Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της νόσου και η αξιολόγηση της ανακοίνωσης του 2009 της Επιτροπής έχει ζωτική σημασία ακριβώς για όλα αυτά που μόλις ακούσαμε από τους συναδέλφους και γιατί δυστυχώς χρειάζεται ακόμη δράση, ακόμη υπολείπονται πολλά. Υπάρχουν πολλά νέα κρούσματα κάθε χρόνο στην Ευρώπη, στον ΕΟΧ, βλέπουμε στην έκθεση του 2010 που μας μιλάει για εκατοντάδες χιλιάδες νέα κρούσματα και πάνω από 100.000 νέα κρούσματα και σίγουρα μπορεί να επιδεινωθεί έτσι περαιτέρω η κατάσταση. Χρειαζόμαστε επενδύσεις, ήδη έχουν γίνει στον τομέα της υγείας, αλλά λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που βιώνουμε αυτή τη στιγμή δυσκολεύουν τα πράγματα. Πρόκειται όμως για τομείς ε, που είναι απαραίτητοι, όπου χρειάζονται επενδύσεις, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και να εκριζώσουμε την νόσο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα θεμελιώδη ρόλο να διαδραματίσει, δηλαδή να πιέζει τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τι απαιτήσει και τα καθήκοντά του στον τομέα αυτό. Επίση, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων διακριτική μεταχείριση ακριβώ λόγω τη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Διακριτική μεταχείριση κατά των εργαζομένων που έχουν χάσει τη δουλειά του ε, ακριβώ επειδή είναι οροθετική. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε μια καθολική πρόσβαση ε, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξαρτήτω ηλικία, ε, φύλου, προέλευση, καταγωγή και ελπίζουμε με την υποστήριξη του Επιτρόπου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο ε, Ρώση, εξ ονόματος της ομάδας της Ευρώπης, της Ελευθερίας και τη Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα για την αντίδραση της Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ω προ την καταπολέμηση της νόσου έχει ήδη υπογραφεί, συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις, αναφέρονται μέσα στο ψήφισμα, παραδείγματο χάρη ο αυξημένος αριθμός νέων κρουσμάτων κάθε χρόνο, 30% των όροθετικών που πάσχουν επίσης από την υπατήτηδα γάμα. Θα πρέπει να συνεχιστεί η εκστρατεία ενημέρωσης για τους κινδύνους μόλυνσης για τον πληθυσμό ε, από αυτήν την νόσο που συνήθως είναι θανατηφόρα ή προκαλεί μεγάλες ε, αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε το αρχικό της ε, κείμενο με μία φράση που φέρει επί της άμβλωσης ε, με την οποία φυσικά διαφωνούμε διότι έτσι αλλάζει η φύση ίδια του ψηφίσματος. Ζητήσαμε κατά τμήματα ψηφοφορία για αυτή την τροπολογία που σχετίζεται με την άμβλωση για να καταργηθεί και έτσι να επανέλθουμε στο αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας βρίσκει σύμφωνους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ψήφισμα για τους πολίτες και κυρίως τους νέους, αλλά δεν θα μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα αν δεν αλλάξει. Τώρα να παρακαλέσω την ε, κυρία Ντότζ από τους μη να πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο αριθμός των ατόμων που ζουν ε, με το AIDS στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ήταν ευξημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος σημαντικά και προβλέπεται ότι θα υπάρξει περαιτέρω έξαρση μέχρι το 2012. Πάρα πολλοί στη χώρα μου ζουν με τον ιό αυτό και έχουμε δύο διαγνώσεις την εβδομάδα για άτομα τα οποία μεταφέρουν το τον ιό ε, και ε, υπάρξει λοιπόν μία αύξηση 20% και η πλειονότητα των περιπτώσεων που διαγνώζονται είναι μεταξύ ανδρών. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα διεθνώς που ζουν και είναι φορείς του ιού ε, εκ των οποίων 2,1 εκατομμύρια παιδιά ε, και που δεν έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία για να με ε, τριάσουν την επέκτασή του. Πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη αντιμετώπιση διότι στιγματίζονται όσοι είναι φορείς και πολλές φορές ε, τα άτομα τα οποία έχουν πληγεί έρχονται για διάγνωση μετά το κρίσιμο στάδιο που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και ε, πολλά από τα άτομα θα μπορούσαν να έχουν ε, εντοπιστεί πιο νωρίς Ευχαριστώ. Εν ονόματι του Συμβουλίου τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Άνταμ Φρόντεκ, ο οποίος ε, είναι υφυπουργό Δημοσίας Υγείας στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη θέση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2011. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αποφέρουν φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του AIDS και εκφράζουν την ε, υποστήριξή τους στους συγγενείς τους αλλά και σε όσους υποφέρουν σήμερα από το AIDS. Σήμερα είναι μια επέτειος. Πριν από 30 χρόνια άρχισε να μαθαίνει ο κόσμος για το AIDS. Οι πρώτες περιπτώσεις εμφανίστηκαν το 1981. Στη συνέχεια πέρασαν 30 χρόνια. 30 χρόνια αγώνα με 30 εκατομμύρια ζωές που χάθηκαν και 16 εκατομμύρια παιδιά έμειναν ορφανά. Ο ιός του AIDS είναι σε πολλές χώρες. 33,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ε, με τον ε, ιό του AIDS και έχουμε 7.000 νέες μολύνσεις κάθε μέρα, ιδιαίτερα στις πιο φτωχές χώρες. Επίσης, είχαμε 30 χρόνια δέσμευσης, συνεργασίας και διαλόγου. Πράγματα που απέβησαν πάρα πολύ σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανθρώπινη εξωπρέπεια είναι και πρέπει να είναι πάντα στο κέντρο ε, του ενδιαφέροντών μας. Έχει υπάρξει πρόοδος και πράγματι έχουν ε, μειωθεί οι μολύνσεις. 19% έχει μειωθεί ο αριθμός των θανάτων στην περίοδο 2004 με 2009. Έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος και στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, στις υποσαχάριες ε, χώρες της Αφρικής για παράδειγμα όπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού ζουν με το AIDS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει στα επιτεύγματα αυτά και είναι περήφανη γι' αυτό και συνεργάστηκε με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, το UNAIDS, την ε, Διεθνή Οργάνωση Υγείας, την UNITAID και άλλους. Το 2010 συνεισέφερε στην καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης, με 53% συνεισφορά στο Ταμείο Global Fund, που ήταν 1.493 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Ήταν το ποσό που δώσανε συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και που μερικές φορές δεν έχουν τα μέσα να δεχτούν τη θεραπεία που τους χρειάζεται. Σε 7 χώρες, 5 από αυτές στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, έχουμε διαπιστώσει μια αύξηση ανάμεσα στο 2001 και το 2009 κατά 25%. Σε συνεργασία όμως με τις χώρες αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί για να αντιστρέψει την τάση. Ζητάει βέβαια περισσότερα προγράμματα πρόληψη και υπηρεσίε τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να απαλληφθεί ο ιός του AIDS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, ε, παίζοντας ηγετικό ρόλο για την αντιμετώπιση του AIDS και ευθυγραμμίζοντας καλύτερα την απάντηση των ευρωπαϊκών θεσμικών ε, οργάνων ε, στα σημερινά πλαίσια, προσαρμόζοντας την αντίδρασή της στα σημερινά πλαίσια όσον αφορά το AIDS. Είναι η πρόκληση μεγάλη, αλλά θέλουμε να σταματήσει η επιδημία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρεται πάντω για την επισκόπηση πρόοδου η οποία περιλαμβάνει τη δέσμευση υπέρ των στόχων της χιλιετίας. Όπως ε, επίσης περιλαμβάνει και τους φιλόδοξους στόχους του 2015 για την απάλληψη του AIDS. έτσι όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το AIDS το 2011 είναι στόχοι που θα μας φέρουν πιο κοντά σε ένα κόσμο χωρίς καθόλου AIDS και χωρίς καθόλου διακρίσεις σε βάρος των θυμάτων του AIDS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνεργάζεται με όσους προσπαθούν να καταπολεμήσουν τον ιό στα πλαίσια της στρατηγικής Getting to Zero, πως θα φτάσουμε σε μηδέν ε, ποσοστά ε, ιού AIDS Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να δουλέψει υπέρ των στόχων του 2015 με 15 εκατομμύρια δηλαδή ανθρώπους που είναι ε, οροθετικοί προκειμένου αυτοί να ε, μπορούν να έχουν θεραπεία με ε, αντιρετροβικά φάρμακα έτσι ώστε να μειωθεί και η μετάδοση της νόσου σε άλλους μέσω σεξουαλικών επαφών ή μέσω ε, ενέσεων που χρησιμοποιούν ε, εκείνοι που παίρνουν ναρκωτικά ή ακόμα και μέσω της μόλυνσης από τη μητέρα ε, που είναι οροθετική στα παιδιά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες γνώσεις που έχουμε όσον αφορά τον ιό και να χρησιμοποιήσουμε την τελευταία λέξη όσον αφορά την πρόληψη και τη θεραπεία. Νέες τεχνολογίες δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα εξαιτία του γεγονότο ότι οι γυναίκε και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτε στον ιό και σε αυτό προστίθενται και οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντε. Οι γυναίκε και τα παιδιά είναι το 50% των ανθρώπων που ζουν με τον ιό του AIDS και είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια σημαντική αιτία και παράγοντα θνησιμότητας στην ε, κατηγορία αυτή ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θέλει να ενισχύσει την δράση της να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία στον παράγοντα του φύλου και να ε, φροντίσει να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για πώς ε, ε, μπορούν να υπάρχουν ασφαλείς επαφές για να αποφευθεί η μόλυνση από τον ιό του AIDS. Άρα χρειάζεται ενημέρωση για τη συμπεριφορά τόσο στις γυναίκες αλλά και όσο και στους άντρες ο πληθυσμός που είναι πιο ευάλωτος, οι άντρες που έχουν σεξ με άντρες δηλαδή, ή κάποιες εθνικές μειονότητες, κρατούμενοι ε, κλπ. Ευάλωτος πληθυσμός πολλές φορές βρίσκεται στο περιφόριο και δεν καταφέρνει να ενημερωθεί καλά-καλά για το πώς μπορεί να προστατευτεί. Ξέρουμε επίσης ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καν πρόσβαση στην ε, ενημέρωση καθόλου. Είναι λοιπόν ζωτική ε, σημασία να έχουν όλοι πρόσβαση σε προγράμματα ενημέρωσης, ε, τεστ για παράδειγμα, εξετάσεις δηλαδή, από τις οποίες θα μάθουν αν είναι οροθετικοί ή όχι, να τους βοηθούμε να μπορούν να χρησιμοποιούν προφυλακτικά είναι αντιμετώπιση δηλαδή που πρέπει να είναι αποτελεσματική. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται ε, σεξουαλικά επίσης, που είναι η, η πατήτιδα Β και Γ για παράδειγμα, η φυματίωση. Θέλουμε λοιπόν ε, προγράμματα για την καταπολέμηση του AIDS να συμπεριληφθούν στα βασικά προγράμματα ε, φροντίδας για την υγεία και στις υπηρεσίες υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι όσοι υποφέρουν από τον ιό του AIDS πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην διαδικασία ε, ελέγχου, πρόληψης και στις πολιτικές στήριξης και στις στρατηγικές και τα προγράμματά μας. Είναι πολύ βασικό να συμμετέχουν και εκείνοι στις προσπάθειές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως εκφράζει την ικανοποίησή της για την σημαντική πρόοδο που έχει ε, μέχρι τώρα επιτευχθεί όσον αφορά την πρόσβαση των ε, οροθετικών σε αντιρετροϊκά φάρμακα. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει μια ανησυχία γιατί σε χώρες πιο φτωχές έχουμε πάνω από 8 εκατομμύρια άτομα τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν τέτοια φάρμακα αλλά δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα τέτοιο πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το έτσι δεν γίνονται ακόμα αρκετά. Εμείς θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε την ένταξη όλων των ατόμων που τα χρειάζονται σαν τη ρετροϊκά φάρμακα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των ε, ατόμων που πλήττονται από τον ιό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρεται πάντως για το γεγονός ότι έχουμε μία μείωση της μόλυνσης από τις μητέρες στα παιδιά είναι κάτι θετικό. Βέβαια θέλουμε να παληθεί πλήρως η μόλυνση των παιδιών από τις μητέρες τους. Οι νέοι, τα παιδιά πρέπει να υποφελούνται από την καλύτερη δυνατόν φροντίδα που μπορεί να υπάρχει ο ιός του AIDS αλλά και άλλες σεξουαλικά μεταδόμενες ασθένειες πρέπει να εντάσσονται και σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο στα προγράμματα καταπολέμησης των ασθενειών αυτών και πρέπει να προστατεύονται οι άνθρωποι που υποφέρουν από το AIDS να προστατεύονται ώστε να μην περιθωριοποιούνται κοινωνικά ούτε να στιγματίζονται μέσα στις κοινωνίες όπου ζουν και να μην υπάρχουν δυσκολίες προκειμένου να εγκαθίστανται σε κάποια χώρα τα άτομα αυτά. Να μην υπάρχει διάκριση κατά των ομοφιλόφιλων και να πάψουν να ισχύουν οι νόμοι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την επιδημία αυτή και ούτε στηρίζουν τις ευάλωτες ομάδες έτσι όπως θα έπρεπε. Σίγουρα βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση, αλλά ίσως ακριβώς γι' αυτό πρέπει ό,τι οι διαθέσιμοι πόροι υπάρχουν να δοθούν για την προώθηση της υγείας. Είμαστε δεσμευμένοι να ενισχύσουμε τα προγράμματα και τον αγώνα γενικότερα που δίνουμε κατά του AIDS και να ενισχύσουμε τα εθνικά συστήματα υγείας και τους πόρους οι οποίοι προσφέρονται στις ε, υπηρεσίες υγείας για να ε, προσφέρεται φροντίδα και θεραπεία στα άτομα που υποφέρουν από το AIDS. Μόνο αν συνεχίσουμε την δουλειά που ήδη κάνουμε, μόνο αν ενισχύσουμε υψηλού επίπεδου παρεμβάσεις και αν κλείσει το χάσμα όπου αυτό υπάρχει σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της και το κάθε κράτος μέλος θα μπορέσουν να ε, μειώσουν τις μολύνσεις από το AIDS, και το στίγμα που βαραίνει πάνω στα άτομα αυτά. Ε, θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον ε, Επίτροπο Ντάλη για τα καταληκτικά του σχόλια και κυρίως για τις ε, δεσμεύσεις της Επιτροπής που περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση για το ηχηρό μήνυμα το οποίο στείλαμε για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά της ασθενείας αυτής του AIDS. Αυτή, αυτό το μήνυμα είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδίως σήμερα διότι λόγω των μέτρων λιτότητος τα οποία έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη πάρα πολλοί πόροι οι οποίοι προηγουμένως είχαν διατεθεί για αυτόν τον τομέα έχουν συρρυκνωθεί τώρα. Και γι' αυτό είναι βασικό το μήνυμά μας σήμερα να είναι ότι μία μείωση του κόστους στις, ε, στους προϋπολογισμούς των χωρών μας ε, πρέπει να τίνει εις ε, την καταπολέμηση της πατάλης και όχι εις την συρρήκνωση των οικονομικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση του AIDS και την έγκαιρη πρόληψη. Κατά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος εις ε, τον αγώνα μας ενάντια αυτής της ασθενείας, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ από το να επιτύχουμε το στόχο μας. δηλαδή να φτάσουμε ένα μηδενικό επίπεδο των μεταδόσεων και των θανάτων αλλά είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε την εργασία αυτή για την επίτευξη των στόχων και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει καταπολέμηση της διακρίσεως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πρόσβαση εις την πρόληψη και στην Ευρώπη και εκτός όπως ελέγχθη από πολλούς από εσά. Δηλαδή χρειάζεται μία μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με ε, το AIDS και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε την εργασία μας στον τομέα αυτό. Ε, υπάρχει μία πλατφόρμα η οποία έχει καταρτιστεί από τα κράτη-μέλη και ε, προσπαθεί να επιβάλλει τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα κράτη-μέλη κατά τρόπον ώστε να υπάρχει συντονισμένη δράση και κατά αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Πολύ, Επίτροπε Ντάλη. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Σας πενθυμίζω ότι το Προεδρείο έχει λάβει μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της ε, συζήτησης και η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι.